Καλησπέρα σε όλους. Αρχίζουμε. Πρώτα με το σημείο 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας το στείλαμε με ηλεκτρονικό τεχειδρομείο Υπάρχει μία αλλαγή μετά από το 15 θα δούμε τα σημεία 17 και 18. Ε, το 16 για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου θα το συζητήσουμε μετά από το σημείο 18. Σημείο 2 ανταλλαγή απόψη ε, ε, των πρακτικών της ε, ΚΟΝΤ σας έχει σταλεί 8 Σεπτεμβρίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Επίσης έχουμε τις 1 Ιουλίου του 2010 και 12 και 13 Ιουλίου που σταλήθηκε στις 15 Ιουλίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνονται. Σημείο 3 έχετε τις διάφορες διαθέσιμες γλώσσες, μετά έχετε και τις κάρτες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, διότι σε λίγο αρχίζει η ψηφοφορία. Για όποιον δεν το ξέρει, η αντιπροσωπεία για την Ουγγαρία 29 και 30 Σεπτεμβρίου έχει αναβληθεί για την επίσκεψη στο ελεγκτικό συνέδριο στις 5 Οκτωβρίου του 2010 θα γίνει το απόγευμα και η ημερήσια διάταξη έχει σταλεί σε όλους στις 20 Σεπτεμβρίου του 2010. Στη συνεδρίαση της 7 Σεπτεμβρίου του 2010 οι συντονιστές ενέκριναν την πρόταση του εισηγητή να γίνει ενημέρωση ε, στις 26 και 27 Οκτωβρίου με παρουσία του ελεγκτικού συνεδρίου και με αντιπροσωπεία του ελεγκτικού συνεδρίου των κάτω χωρών και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Αυτή η συνεδρία αναβάλλεται για τις 15 Νοεμβρίου του 2010 διότι δεν μπορεί να είναι παρόν το ελεγκτικό συνέδριο. Καλωσορίζουμε ορίζουμε την κυρία Μπόλντι, την κυρία Κόβα και την κυρία Σιράλτο που είναι τα νέα μέλη της γραμματείας. Λοιπόν, όλοι σας έχετε την κάρτα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και προχωρούμε στην ψηφοφορία των σημείων 4, 5, 6, 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης. Πρώτα ψηφίζουμε το σημείο 4 δύο οργανική συμφωνία σχετικά με τη συνεργασία για θέματα προϋπολογισμού. Ψηφίζουμε συνολικά τη γνωμοδότηση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Okay. μου είπαν να περιμένω γιατί όπου να είναι έρχονται οι, οι κάρτες για τους ξεχασιάριδες συναδέλφους. Aspettiamo qualche minuto. Ma lui pure manca. Sì, questi due, Pancit e Corsolino e Deutsch manca. Lo facciamo forse con, con mano. Sì. Vabbè, cominciamo, facciamo una cosa, facciamo per chi non ha la carta. Κοιτάστε, όποιος δεν έχει την ηλεκτρονική του κάρτα, σηκώσει το χέρι του. Και οι υπόλοιποι με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Στο 19.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 Vado. Ok. Passiamo adesso alla votazione del punto. Yes. Okay. Ehm, Presidente, ich muss. Ehm, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ε, να, να, να κάνω μία επεξήγηση ψήφου για να εξηγήσω και την θέση των σοσιαλδημοκρατών για την τροπολογία 2 σχετικά με την έκθεση του κυρίου Μπαλσίτης. Εμείς αύριο θα ψηφίσουμε, σε κοινή ψηφοφορία, με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Η ομάδα εργασίας για τον προϋπολογισμό της σοσιαλιστικής ομάδας θεωρεί ότι, ότι υπάρχει ρίσκο αντίφασης με αυτήν την τροπολογία και την αποσύραμε. Ο κύριος Μπαλσίτης το δέχτηκε, οπότε δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε γιατί αποσύρθηκε. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις, ας πάμε στο σημείο 5 σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθμός 6 2010 στον γενικό προϋπολογισμό του 2010 Δεύτερο τμήμα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο, τμήμα 3 Επιτροπή, τμήμα 10 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. 22 υπέρ. Η 2 αποσύρθηκε. Τροπολογία 3. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 16 υπέρ 2 κατά 5 αποχές το ψήφισμα στο σύνολό του αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίες 21 ψήφι υπέρ, ένας κατά και μία αποχή. Passiamo adesso al punto 6 dell'ordine del giorno. Σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη. τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των κοινοτήτων. Η εισηγήτρια έχει το λόγο. Γιατί... η ρελατούρε. Η κυρία Χέρτζοκ. Thanks very much, Chairman. I... Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συνεισηγητές και συνεισηγήτριες. Τρία στοιχεία θα ήθελα να τονίσω. Θα ζητήσουμε ίση μεταχείριση και διαφανέστατες διαδικασίες για όλους και όλες. Για μας είναι σημαντικό οι πειθαρχικές διαδικασίες να συμφωνούν με όλα όσα έχουμε πει στο παρελθόν. Θα ήθελα δε να τονίσω ότι αποσύρω τις τροπολογίες 11 και 12. Δεν φαντάζομαι να υπάρχει πρόβλημα και νομίζω ότι μπορούμε τις υπόλοιπες να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Αλλιώς μία-μία. Τέλος πάντων, οι 11 και οι 12 αποσύρονται. Σύρονται. Λοιπόν, εγώ αρχίζω την ψηφοφορία ψηφίζοντα κανονικά, χωρί ε, ψηφοφορία μπλοκ για να μην μπλεχτούμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 1, αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22 υπέρ, 4 κατά. Τροπολογία 2, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 22-4. Μία αποχή. Τροπολογία 3. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 21 4 και μία αποχή. Τροπολογία 4. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 25 υπέρ και μία αποχή τροπολογία 5 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 25-2 τροπολογία 6 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 26 υπέρ και μία αποχή Τροπολογία 7. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 24 υπέρ 3 κατά. Τροπολογία 8 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 27 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 9 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 23-3. Τροπολογία 10. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 11 και 12 έχουν αποσυρθεί. Τροπολογία 13 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 27 ψήφι υπέρ. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση στο σύνολό της, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 25 ψήφοι υπέρ και 2 ψήφοι κατά. Ψηφίζουμε το, ε, προχωράμε στο σημείο 7 γνωμοδότηση για τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο Τρίτο Τμήμα Κομισιόν. Εάν δεν υπάρχουν τοποθετήσει, αρχίζουμε. Τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 12-15. Λοιπόν, τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι πέρα, 6 κατά. Τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίας. Εγκρίνεται 22 υπέρ 5 κατά τροπολογία 5 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 25-2. Τροπολογία 6 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 26 υπέρ ένας κατά ψηφίζουμε το ψήφισμα συνολικά αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται υπέρ ένας κατά και μία αποχή σημείο 8 είναι η το δεύτερο σχέδιο για την απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το 2008. Η κυρία Ματιούθελ, το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6 και ευχαριστώ τους και όδης το ελεγκτικό συνέδριο, τη γραμματεία διότι μετά από ένα χρόνο ε, δουλειά έρχεται και πάλι η έκθεση στην Επιτροπή μας και μετά από τόση δουλειά καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό που ικανοποιεί τους πάντες. Grazie, procediamo quindi alla... Mm, Ψηφίζουμε. Και αρχίζουμε με την πρόταση απόφαση στο σύνολό της αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Έχουμε ένα ΕΛΚ παραπανίσιο. Ξαναψηφίζουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. 26 ψήφισαν, κανένας δεν καταψήφισε. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση απόφαση στο σύνολό τη. Σημείο 2 για το κλείσιμο των λογαριασμών. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Πάμε τώρα στο σχέδιο ψηφίσματος. Τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 25 ψήφοι υπέρ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Οι πέντε, εμείς ως ομάδα είμαστε υπέρ αυτού που λέει, αλλά ως προσθήκη, όχι αντικατάσταση του αρχικού κειμένου. Μήπως οι κύριοι Σταυρακάκης και Γκάγερ θα μπορούσαν να εγκρίνουν αυτό το αίτημα για προσθήκη. Ναι, άμα Σύμφωνο από το νεύμα που μου έγινε. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Η τροπολογία 5 παράγραφος 4. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 16 ψήφοι υπέρ, 10 κατά και μία αποχή. Ποιος ήθελε το λόγο? Α, για την παράγραφο 6 μάλιστα. Θέλαμε να διαγράψουμε το όνομα του νέου διευθυντή στην παράγραφο 6. Θεωρεί ότι ο νέος διευθυντής του κολεγίου, διαγράφουμε, θα παρουσιάσει και τα χωρίς να λέμε όνομα. Αρχίζει η ψηφοφορία της τροπολογίας 6. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 26 υπέρ μια αποχή 7 αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 16 ψήφοι κατά και 10 ψήφοι υπέρ τροπολογία 8 αρχίζει ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26-1. Τροπολογία 10. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 18 κατά 9 υπέρ. Τροπολογία 11. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. Ψηφίζουμε στο σύνολό του το ψήφισμα, όπως τροποποιήθηκε και αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Ετήσια έκθεση 2010 της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. Την παρουσίαση θα κάνει ο διευθυντής της Όλαφ, ο προσωρινός διευθυντής, ο ο Νίκολας Ήλετ και του δίνω το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Κατά διάφορα της συνολικής διάρκειας, η οποία καλύπτεται από την έκθεση δραστηριοτήτων, δηλαδή το 2009, ε, ηγείται ο Hans Hermann Brunner της Όλαφ. Υπό τη δική του ηγεσία η Όλαφ σε όλους τους μίσους της εντολής ε, πέτυχε μεγάλες επιτυχίες. Θα ήθελα εδώ παραδειγματικά να αναφερθώ σε κάποιες επιτυχίες μόνο. Εσωτερικές, ε, εσωτερική έλεγχη στα θεσμικά όργανα. αλληλετική έλεγχη και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες σε τομείς που αρχικά δεν καλύπτονται καθόλου. Συντονισμός των ελληνικών δράσεων. Περιορισμός ε, του λαθρεμπορίου ε, τσιγάρων με διάφορα μέτρα, παραδείγματο χάρη την σύναψη συμφωνιών με τους μεγαλύτερους παραγωγούς. Και μόλις σήμερα το πρωί υπέγραψα μια τέτοια συμφωνία ακόμα. Ένωνες ε, προσπάθειες στα νέα κράτη-μέλη στις υποψήφιες χώρες και στις χώρες της, Επιτρο... της Ευρωπαϊκής Πολιτικής ειδικό ρόλο στην καταπολέμηση των απατών σε σχέση με σχέδια αναπτυξιακής βοήθειας, στη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνούς οργανισμούς και σε, με άμεση συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική. Ο τρόπος με τον οποίο η Όλαφ αναπτύχθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια και πώς προασπίζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παραδειγματικός σε διεθνές επίπεδο. Με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε θα περάσω τώρα στα αγγλικά. και θα παρουσιάσω τα κύρια σημεία της 10ης έκθεσης δραστηριοτήτων του Όλαφ, δίνοντάς μια συνεργική εικόνα των βασικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του 2009. Σε ελληνικέ γραμμέ το 2009 ήταν ένα έτος συνεχής και παγίωση 10 χρόνια μετά την ίδρυση της Όλαφ. Ο όγκος πληροφοριών που λάβαμε αυξήθηκε από 802 νέα στοιχεία το 2005 σε 969 το 2009. Ναι. Πέρσι πήραμε 740 αποφάσεις σε σχέση με νέες ε, πληροφορίες που λαμβάνουμε. Από τις 740 αυτές αποφάσεις, οι 220 οδήγησαν στο άνοιγμα μιας υπόθεσης, δηλαδή κάπως περισσότερες από τις 204 που είχαμε το 2008. Από τις 220 αυτές υποθέσεις που άνοιξαν, μπορέσαμε 148 να πραγματοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι και οι υπόλοιπες 72 ήταν υποθέσεις συνεργασίας ή ενίσχυσης. Από τις 148 υποθέσεις που διερευκάναμε εμείς, η 99 ήταν εσωτερική έλεγχη και 49 εσωτερική. Θα ήθελα να σας αναφέρω τους τομείς στους, του προπολογισμού στους οποίους έκανε αυτές τις έρευνες η ΟΛΑΦ. Σε ποσοστά. 33% ήταν μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. 18% στη Γεωργία, 13% στην εξωτερική βοήθεια, 11% στις άμενες δαπάνες, άλλες όπως ορίζονται από την Κομισιόν, 10% διορθωτικά ταμεία, 10% στη τελωνία και 5% για τα τσιγάρα. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλη του 2009 είχε η ΟΛΑΦ 369 ενεργές έρευνες, 354 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 15 σε υποψήφιες χώρες. Η ετήσια έκραση δίνει μια σύντομη περιγραφή ορισμένων από τις υποθέσεις αυτές στους διάφορους τομείς. Όπως καταλαβαίνετε όμως, για νομικούς ε, ε, πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ επιβλεκτικοί όσον αφορά τις λεπτομέρειες που υποβάλλουμε. Πιο επιβλεκτικοί κάθε χρονιά. Αλλά θα είμαστε κατανοτών ανοιχτοί δίνοντα απαντήσει που ίσως θέλετε να λάβετε. Τα τέλη του 2009 είχαμε καλέψει 250 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είχαν ανακληθεί σαν αποτέλεσμα των δράσεων που ολοκληρώσε η Όλαφ. Τα αποτελέσματα αυτά διακυμαίνονται πολύ από χρόνο σε χρόνο, γιατί σε ορισμένα χρόνια υπάρχουν πάρα πολλοί ψηλά ποσά. Παραδείγματο, το 2009, μία και μοναδική περίπτωση στην Ιωργία αφορούσε 113 εκατομμύρια, τα οποία ανακτήθησαν. Mm. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε τέσσερι τομεί των δραστηριοτήτων τη Όλαφ, οι οποίε δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην τρέχουσα έκθεση. Πρώτον, η πολιτική της Όλαφ είναι να εξετάζει όσο περισσότερο όσο πάει και περισσότερο σοβαρές υποθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι ασχολούμεθα μόνο με τις πιο σοβαρές υποθέσεις, ασχολούμεθα και με λιγότερο σοβαρές, αλλά όπου είναι δυνατόν ασχολούμεθα με τις πιο σοβαρές. Κάναμε περαιτέρω πρόοδο επίσης στις διαδικαστικές ε, τυχές ε, των εργασιών μας. Εισάγαμε μια πολιτική de minimis, ούτως ώστε η Όλαφ να μπορεί να χρησιμοποιεί τους πόρους πιο αποτελεσματικά και να ε, συγκεντρώνει την προσοχή του σε επιπεθώσεις που προσφέρουν μια σαφή προστιθέμενη αξία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ενδεικτικά ε, οικονομικά κατόφια για τη λειτουργία των ερευνών όλα στους διάφορους τομείς. Και όταν οι περιπτώσεις αυτές δεν φτάνουν το εν λόγω ε, κατόφλι, αναφερόμαστε σε άλλες υπηρεσίες, όσο παραδείγματος στην υπηρεσία των της Κομισιόν. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτή η προσαρμογή της πολιτικής μας εξακολουθεί να είναι ευθυγραμμισμένη με την πολιτική μηδέν ανοχής που έχει υιοθετηθεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισαγάγαμε νέες διαδικασίες ακολουθήσεις ε, για να εξετάζονται οι αρμοδιότητες ΟΛΑΦ σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν και τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη συνοχή που δίνεται στις περιπτώσεις που εξετάζουμε. Επίσης, εφόσον μπορούσαμε, ε, κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες ε, εκτιμήσεις των οικονομικών απολειών που προλαμβάνονται από τις δράσεις μας. Ένα νέο εγχειρίδιο της Όλαφ εισήχθη τα τέλη του 2009. Και αυτό ήταν το τελευταίο επίσημο έγγραφο που υπέγραψε ο κύριος Μπρουνέρ. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εργασία μας βασίζεται στο κράτος δικαίου και στο να μην λαμβάνουμε την, ε, να μην προασπίζουμε τα συμφέροντα των μεν ή των δε. Έχουμε προχωρήσει από μια κατάσταση στην οποία ο στόχος μας ήταν να είμαστε λογικοί και δίκαιοι στο διοικητικό ε, νομικό τομέα που τώρα που σεβόμαστε όλες τις δικαστικές ε, ε, διαδικασίες. Είμαστε πολύ πιο αυστηροί και οριστικοί στις διαδικασίες που ακολουθούμε. Δεύτερον, τονίζουμε ιδιαίτερα την πρόληψη των ε, απατών και την ανάλυση μια κοινή στρατηγική πρόληψη των απατών για τα διαδοτικά ταμεία υιοθετήθηκε ή εφαρμόζεται από την ΟΛΑΦ σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση και Περιφερειακή Ανάπτυξη και έχει σαν στόχο να γίνουν καλύτερα κατανοητικέ οι διαδικασίε αυτέ πρόληψη των απατών από, τα... από τι άλλε υπηρεσίε και γενικέ διευθύνσει τη και από τα κράτη-μέλη. Δίνουμε επίσης αναλυτική ενίσχυση σε στρατηγικά, τακτικά και λειτουργικά επίπεδα σε άλλες υπηρεσίες της Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Ο στόχος πάλι είναι να αυξηθεί η κατανόηση των ε, υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τα οικονομικά όσον αφορά ποιε είναι οι συνήθεις ατασταλίες και ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι απάτε. Ένα τρίτο τομέα, στον οποίο θα να στην προσοχή σα, κύριε Πρόεδρε, στον οποίο δράσαμε ιδιαίτερα, ήταν μέσα στα πλαίσια των εξωτερικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τώρα μια ειδική μονάδα, εδώ και αρκετά χρόνια, για τις έρευνες της υπηρεσίας αυτές. Όπως γνωρίζει πολύ καλά η υπηρεσία σας, αυτό είναι τομέας υψηλού κινδύνου για κακή διαχείριση, για απάτη και διαφορά. Η Όλαφ μπόρεσε να βρει μια σειρά τομέων όπου υπάρχουν έντονοι κίνδυνοι και που τώρα μπορούν να αντιμετωπιστούν με συνεχή και εις βάθος συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τέλος θα περάσω στον τομέα εισο... εσόδων συγγνώμη, του προπολισμού που πολλές φορές παραβλέπουμε, που είναι όμως επίσης σημαντικό. Η κοινή ε, ε, πράξη ε, τελωνίων, διάβολο 2, που οργανώσει ο ΛΑΦ Ένωση 45 μέλη της ΑΣΕΜ που ενώνει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις περισσότερες χώρες της Ασίας για να το καταπολεμηθεί το εμπόριο σε πλαστογραφημένα αγαθά. Αυτό οδήγησε στην ε, κατάσχεση 65 εκατομμυρίων τσιγάρων και 369.000 άλλων παραποιημένων ε, αγαθών. Ο ρόλος ε, της ΟΛΑΦ εδώ ήταν το ρόλο του συντονιστή. Τα κύρια στοιχεία ήταν μια πλατφόρμα ε, πληροφορικής μας επέτρεψε σε πραγματικό χρόνο συνεργασία και ανταλλαγή ε, πληροφοριών βασιζόμενοι σε μια δυνατότητα που έχουμε στο υπόγειό μας και που οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτό θα είναι πολύ χαρούμενοι να μπορούν να σας το δείξουν. και που καταπολεμά ένα μεγάλο ποσοστό του λειτουργικού μας προϋπολογισμού. Έχουμε αυτή τη πλατφόρμα που μπορεί πραγματικά όταν χρησιμοποιηθεί να πετύχει αυτά τα καταπληκτικά αποτελέσματα στις υπηρεσίες τελωνίων όχι μόνο των κρατών μελών αλλά και οποιασδήποτε τρίτης χώρες που θέλουμε να εντάξουμε μέσα στο... στις προσπάθειές μας. Και εδώ αναφέρθηκα στην διεθνή συνεργασία και θέλω να τονίσω τον ρόλο που παίζει όλα αυτά τώρα μέσα στα πλαίσια των διεθνών οργανώσεων που ε, δρούν ενεργά για την καταβαλώμηση της διαφθοράς και της απάτης στα σχέδια ενίσχυσης και ανάπτυξης. Προσπαθούμε να εργαστούμε και συνεργασία και με άλλες ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την Europe Aid Cooperation Office, και το την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπηρεσιών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ΕΚΟ δηλαδή. Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, έχω να παρατηρήσω τρία πράγματα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ε, πω που επαναλαμβάνουμε πάντα πάντα στην Όλαφ κάθε φορά που υποδεχόμαστε νέα μέλη στην Όλαφ ότι εμείς στην υπηρεσία μας είμαστε επιβεβαιωμένοι ότι καμιά δουλειά στην, Ευρω... Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σημαντικότερη από εκείνη που κάνουμε εμείς. Άλλες πολιτικές έχουν ένα πιο έντονο προφίλ, νομισματική ένωση, η νέα αγορά, όλα αυτά τα μεγάλα σχέδια τα οποία είναι γνωστά και που δείξαν στη σημερινή, στο σημερινό επίπεδο ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Εμείς όμως έχουμε την τιμή να κάνουμε ένα έργο το οποίο αμήνεται της ε, ε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, ξέρουμε ότι βέβαια και εμεί υποκείμεθα στις πιέσεις που ε, όσο πάει και περισσότερο ε, επιβάλλονται στις ε, δημόσιε υπηρεσίε και σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πίεση αυτή των πόρων μας κάνει να αναγκαζόμαστε να επανεξετάσουμε τις προτεραιότητες μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μελλοντικέ απειλές. Το προσωπικό μας κατανοεί την ανάγκη αλλαγής και χαίρονται για τις προσκλήσεις που υπάρχουν. Παραμένει όμως σημαντικό στην πολιτική διαδικασία να εξακολουθεί να διατηρήσει την ανεξαρτησία και την απολυσματικότητα μιας λειτουργικής υπηρεσίας και επίσης όσον αφορά το ηθικό του προσωπικού. Κύριε Πρόεδρε, εξ αρχή έχουμε συνεργαστεί έντονα με την δική σα ε, επιτροπή που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Αυτή η εμπιστοσύνη που μα δείχνετε ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη ευσία για μα. Το τελευταίο θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτσεβιτ ζήτησε το λόγο. Α? Πρόεδρε. Χαιρόμαστε που οι δραστηριότητε τη αυτό το 2009 ε, ήταν τόσο πιο αποτελεσματικέ και μπόρεσαν να αναπτύξουν τέτοια τεράστια ποσά ευρώ για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθούμε όμως να έχουμε προβλήματα στα κράτη-μέλη. Ένα από αυτά είναι η ανταλλαγή των στοιχείων. Στην Λιθουανία αυτή τη στιγμή έχουμε πέντε υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με το θέμα των ε, οικονομικών εγκλημάτων και τη διαφορά. Αλλά δεν θέλουν να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους. ίσως είναι καλύτερο να υπάρχει ένα συγκεντρωτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Όλαφ και να υπάρχει μια υπηρεσία που είναι αρμόδια για την αλληλεγγύη αυτών των, των πληροφοριών. Ο αριθμό ε, των υποθέσεων που εξετάστηκαν ε, κατά τη διάρκεια του 2009 να ολοκληρωθείς που ολοκληρώθηκαν δεν ήταν πια 65% ήταν 55% και θα πρέπει να γίνει να έχουμε και εδώ κάποια πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα για το σημείο 2 που αφορά λέει διάφορες χώρες και τον αριθμό των ερευνών που έχουν γίνει σε αυτές. Κατανοώ ότι υπάρχουν αμφιβολίες χρειάζεται φρόνηση γιατί είναι προφανές ότι αν δεν υπάρχουν φάκελοι για ορισμένες χώρες αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν ενδιαφέρεται το κράτος να συνεργαστεί με την Όλαφ. Ίσως η Δανία και η Φιλανδία να μην έχουν καμία υπόθεση. Αλλά Φαντάζομαι ότι όταν γίνεται μια αποτίμηση αυτών των στατιστικών στοιχείων ότι θα μπορούσαμε να δούμε ποιες χώρες είναι οι πιο προβληματικές. Πού αντιμετωπίσατε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί οι αριθμοί κάθε αυτούς δεν είναι πολύ αποκαλυπτικοί. Μπορεί να αφορούν διάφορες καταστάσεις και διαφορετικού βάρους. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν μπορείτε να κάνετε μια αποτίμηση πιο σε βάθος. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγγνώμη κύριε Ελέτ, θα ήθελα να εκφράσω σε συγχαρητήριά μου στην ΟΛΕΦ για την εργασία που έχει επιτελέσει, για το έργο που έχει επιτελέσει. Η έκθεση αυτή πραγματικά αποτελεί ένα τεράστιο κβαντικό άλμα σε σχέση με την περασμένη έκθεση ίσως οι συνάδελφοι δεν έχουν παρακολουθήσει τόσο στενά τις εξελίξεις, δεν το ξέρουν, ναι, αλλά εγώ ασχολήθηκα ε, έντονα με το θέμα και γι' αυτό πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει βελτίωση της παρουσίασης. Ταυτόχρονα, και αυτή είναι η πρώτη μου ε, ερώτηση, υπάρχει προσπάθεια μιας ε, νέας ονοματολογίας. Το να έχουμε έναν ορισμό του τι είναι απάτη αλλά υπάρχει για πρώτη φορά μια προσπάθεια ποσοτικής αξιολόγησης του απατών. Δηλαδή πόσο ποσοστό του κυρωτικού προπολογισμού ε, είναι αντικείμενο ίσως απατών. Καλό είναι αυτό, ευχάριστο είναι, χρήσιμο είναι, αλλά υπάρχει μια φαιά ζώνη πολύ μεγάλα. Εγώ καταλαβαίνω συζήτηση το υπέρ και τα κατά, το πόσο Σήμο είναι αυτό και πως όχι. Η έκθεση είναι πραγματικά πάρα πολύ προσεκτική. Μπορούμε πολλά να κάνουμε τα στοιχεία που μας δίνει, αλλά βλέπω να υπάρχει τελικά μία προσπάθεια ε, αν θέλετε, για την κακή διαχείριση και για το ακόμα και για γραμματικότητα Ποιος είχε την ιδέα για την στατιστική αυτή καινοτομία. Δεύτερον, αυτό είναι μια έκθεση της Κομισιόν. Υπάρχει και έκθεση Σόλαφ όλα αυτή την εργασία της, αλλά αυτή είναι η έκθεση Γενικής Γραμματείας. Δεν με ενδιαφέρει μονάχα ποιο ε, όρισε τους τίτλους, αλλά πόσο μεγάλη ήταν η επίδραση του, της Όλαφ. Ποια είναι η δική σας άποψη για τις ε, καινοτομίε αυτές που έχουν εισαχθεί. Αυτά είναι δεύτερη ερώτηση. Τρίτη ερώτηση αφορά μια από τι κύριε βελτιώσεις. Δηλαδή τη βελτίωση της, ε, των δηλώσεων για ε, περιπτώσεις υποψίας απατών. Εδώ είχαμε, δεν ξέρω, θυμάμαι πόσες, 100, ε, 200, δεν θυμάμαι και τώρα έχουμε 800 περιπτώσεις. Παραδείγματο το αγροτικό τομέα αυξήθηκε κατά 43% το ποσοστό αυτό. Οι δηλώσεις δηλαδή υποψίας απάτης. Και για το μέλλον πώς αξιολογείται αυτό το σύστημα και πώς θα το επιβάλλετε. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι καλό το σύστημα αυτό. Και όσο πιο ευρέως χρησιμοποιηθεί και από τους χρήστες, θα μπορέσουμε περισσότερο να έχουμε δηλώσει αυτές υποψίες και θέλουμε πραγματικά οι περιπτώσεις απάτης να δηλώνονται. Και συμφωνώ με αυτό που είπατε για τη μηδενική ανοχή. Η επόμενη μου ερώτηση αφορά ένα σκοτεινό κεφάλαιο. Δηλαδή την ε, ανάκτηση των ποσών αυτών. Αναφέρεται αναλυτικά και πολύ ωραία. Είμαι πολύ ευγνώμων για την πληροφορία αυτή. των αγροτικών με παραδείγματος 50 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορούν να ανακτηθούν. Γενικά 1,36 δισεκατομμύρια. Και ανακτήθησαν 167 εκατομμύρια, δηλαδή κάτι παραπάνω από 10%. Ποια είναι τα προβλήματα μέτρα για να αυξηθεί το ποσοστό αυτό. Και μετά έχω μια ερώτηση για την αγαπητή μας χώρα μέλος, την Ιταλία. Στην Ιταλία, ναι. Αναφέρεται ότι από το 2004, για το 2004 που ολοκληρώθηκε τον οργανισμό, το 60% των ε, περιπτώσεων ε, απάτης αφορούν την Ιταλία. Το 60% για το 2004. Πώς προβλέπετε τη συνεργασία με τη χώρα αυτή Πώς θα, επίσης ξέρουμε ότι η ενάκτηση των όποσων αυτών είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά το θέμα. Αυτές οι ερωτήσεις και σας ευχαριστώ πολύ. Ähm, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω τέσσερις ε, να σας στον κύριο Άιλετ. Ε, Συμφωνώ και εγώ με την ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε όσον αφορά τις ε, υποψίες απατών στην Ιταλία. Και από ό,τι διάβασα στην περίληψη, το μόνο που μπορούσα να μελετήσω μέχρι στιγμής, βλέπω ότι υπάρχει και ένας άλλος ε, τομέας όσον αφορά τα Βαλκάνια και μελλοντικά μάλιστα τα Δυτικά Βαλκάνια. Τα τους τελευταίους 12 μήνες τι έκανε κυρίως η Όλαφ για να μπορέσει να αντιδράσει στους κινδύνους και τις απάτες στα Βαλκάνια. Δεύτερη ερώτηση. Όταν πρόκειται για διεθνή συνεργασία, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η Όλαφ στο μέλλον θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Διεθνή Ακαδημία Καταπολέμησης Απάτης που έχει έδρα αυτή τη στιγμή στην Βιέννη. Τρίτο σημείο. Η συνεργασία ε, μεταξύ Όλαφ και Eurojust. Πώς λειτουργεί και πώς θα ε, σχηματιστεί στο μέλλον. Και το τέταρτο σημείο αφορά τον αριθμό των ερευνητών. υπάρχει εδώ ένας αριθμός για investigators και operators. Ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων αυτών, των ερευνητών επιτόπου, ποιος είναι. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο μέσα στον κύριο Άλεπ να απαντήσει. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. πολύ ευρύ το φάσμα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω, αλλά αν έχετε συμπληρωματικές, να τις θέσετε και αυτές. Για την ανταλλαγή των δεδομένων. Εμείς μιλάμε για θέματα προστασίας τους πάρα πολύ. Συνήθως όταν δεν ανταλλάσσονται τα δεδομένα, ενώ θα έπρεπε, ο λόγος δεν είναι ότι δεν υπήρχε αρκετή, ότι εμποδίστηκε η ανταλλαγή από την πολιτική προστασία, αλλά ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά η διαδικασία αυτή, διότι οι μηχανισμοί προστασίας δεδομένων επιτρέπουν την ανταλλαγή τους, εφόσον είναι βεβαίως δικαιολογημένοι Από ό,τι όμως ξέρουμε το καλύτερο είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μάλλον παρά να εφαρμόζονται νέοι μηχανισμοί τελείως. Θα ήθελα τώρα να σχολιάσω αυτή τη φιλοδοξότατη πρόταση που έγινε για μια νέα υπηρεσία προστασίας των δεδομένων. Αυτή είναι αμφιλεγόμενη ιδέα Εμένα θα μου διευκόλυνε τα πράγματα, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Και τέλος, τέλος, τέλος για τον πρώτο μιλητή δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ρωτούσε γιατί ο αριθμός των υποθέσεων που δεν, όπου δεν δόθηκε συνέχεια έπεσε από 65 σε 55% από το 8 στο 9 και η απάντηση είναι ότι στη φάση αυτή δεν είμαστε βέβαιοι αν έχει αν είναι παγιωμένη αυτή η κατάσταση και τάση. Προς στιγμή θα έλεγα ότι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είμαστε πιο συγκεκριμένοι με βάση μόλις τα δεδομένα ενός χρόνου. Δεύτερον, ή μάλλον πρώτη ερώτηση του δεύτερου ομιλητή. Ποιες χώρες μπορεί να είναι οι πιο δύσκολες από άλλες, πιο δύσκολες από άλλες. Είναι προφανές ότι τα προβλήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Μεταξύ άλλων και για λόγους ιστορικούς, θεσμικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικού, δομικούς κτλ. Το σημαντικό νομίζω είναι να δεχτούμε ότι απλώς και μόνο επειδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε μια χώρα δεν σημαίνει ότι η χώρα αυτή είναι αναγκαστικά προβληματική. Ίσως να ήταν εάν η κατάστασή της ήταν χειρότερη από αλλονών. Αλλά θα μπορούσε αυτό και να δείχνει απλώς ότι έχει επιδείξει μεγαλύτερη συνεργασία με εμάς ή ότι πολλές περιπτώσεις συνδέονται μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη στη Βολγαρία συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πολλές περιπτώσεις αλλά παρόμοιες όλες μεταξύ τους. Παρόμοιες απάτες. Εγώ δεν νομίζω ότι η δουλειά μου είναι να ονοματίσω εδώ ποιες μεμονωμένες χώρες μέλη είναι προβληματικές. Αυτό αφορά καλύτερη λειτουργία του δικαστικού συστήματος και των υπηρεσιών γενικότερα, ιδιαίτερα σε νεότερες χώρες μέλη, αλλά υπάρχει και το θέμα, το θέμα υπάρχει και σε παλαιότερες χώρες μέλη. Και εγώ είμαι πολίτης μιας νεότερης χώρας μέλους. αλλά όσο και να εξετάσω το παρελθόν πάλι βρίσκω ότι μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις στην καλύτερη δημόσια διοίκηση και καταπολέμηση των ατών. Υπάρχουν και ιδιαιτερότητες όπως ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι γίνονται στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο επειδή εκεί εδρεύουν τα όργανα και εκεί επομένως εξετάζονται, γίνονται και οι περισσότερες απάτες. Αλλά άμα δούμε τους αριθμούς πιο λεπτομεριακά θα καταλάβουμε ότι σε μερικές χώρες μέλη υπάρχει περισσότερη συνεργασία και περισσότερες υποθέσεις σε σύγκριση με τον πληθυσμό τους αλλά και με τις δαπάνες στις χώρες αυτές. Το να πούμε ότι υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις στη Γερμανία από όπου αλλού δεν λέει και πολλά. Λόγω του μεγέθους της Γερμανίας και του ύψους του προϋπολογισμού που δαπανάται εκεί. Δύο από τις μεγαλύτερες χώρες μέλη, εξών και η δική μου μαζί με μια γειτονική, έχουν λιγότερες, λιγότερους ελέγχους εκθέσεις και άρα και λιγότερες περιπτώσεις. Και εδώ δεν κρίνω κατά πόσον αυτό δείχνει ότι τα πράγματα είναι σοβαρά ή όχι είναι ένα απλό γεγονός στατιστικό τώρα το ερώτημα της δοκτορέσης Γκρέσλε την ευχαριστώ για όσα ευγενικά είπε για τις προσπάθειές μας βελτίωσης της δόμησης του κειμένου Το ποιο είναι το ακριβές επίπεδο απάτης είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Δεν προσπαθήσαμε να το βάλουμε σε αριθμούς αυτό. Γιατί κάναμε προσπάθειες αλλά καταλήξαμε ότι δεν υπήρχε καμία αξιόπιστη μέθοδος για να μπορέσουμε να προβλέψουμε απάτες. Ξέρουμε ποιες απάτες έχουν ταυτιστεί ως τη, οι λιγότερο πιθανές, όχι ως οι περισσότερο πιθανές, από τις χώρες μέλη όταν υποβάλλουν τις εκθέσεις τους. Και σε αυτήν τη βάση γράφτηκαν, αναφέρθηκαν οι αριθμοί που εμφαίνονται στην έκθεση της Όλαφ. Στην έκθεση όμως της Επιτροπής της Κομισιόν, αύριο, θα δείτε πιο λεπτομερή στοιχεία που βασίζονται όμως σε όσα υπέβαλαν οι χώρες μέλη. Η έκθεση της Κομισιόν για την απάτη ή για τις απάτες σύμφωνα με το 325 που θα συζητήσετε αύριο συνετάχθη σε συνεργασία με την Όλαφ, όχι όμως αποκλειστικά από την Όλαφ. Και η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών και άλλες συνεργάστηκαν. Η διαφορά είναι ότι καλύπτει όλες τις δικαιοδοσίες της Κομισιόν εκείνη και βασίζεται σε αριθμούς όπως είπα και πριν που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη και με βάση την γνωστή διαδικασία για τις δημοσιεύσεις της Κομισιόν ενώ η δική μας έκθεση δραστηριοτήτων της Όλαφου συζητάτε σήμερα, συνετάχθη από, τη Γενική, το Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, με δική του ευθύνη και βασίζεται στις ανεξάρτητες τις δραστηριότητες που δεν διαχωρίζονται βέβαια απόλυτα και από τις υπόλοιπες Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ της δικής μας έκθεσης και της έκθεσης της Κομισιόν. Οι ατασταλίες τώρα επηρεάζονται από τους ορισμούς και την πρακτική που μπορεί να αλλάζουν. υπάρχει το σύστημα επιτήρησης ατασταλιών ΣΕΑ και γενικότερα θα ήθελα να σας πω και να σας μεταφέρω ως μήνυμα ότι δεν, ε, δεν παίρνει τα χρήματα τις επιστροφές η Όλαφ η ίδια αλλά τα κράτη. Εμείς απλώς προσπαθούμε να ταυτίσουμε σε ποιες περιπτώσεις υπάρχουν στοιχεία που οδηγούν σε απόφαση επιστροφής χρημάτων. Αποζημίωσης ή επιστροφής. Πρέπει είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε ακριβώς ποιος κάνει τι, αλλά βασικά δεν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για τις επιστροφές, αλλά άλλοι, στους οποίους εμείς δίνουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εισπράξουν Τέλος, για την Ιταλία. Στη σχέση μας με την Ιταλία έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Οι Ιταλοί έχουν δημοσιονομική αστυνομία, πράγμα που δεν διαθέτουν άλλες χώρες. Έχουν πολλούς πόρους για την καταπολέμηση των απατών αυτών και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων το δικαστικό τους σύστημα είναι πολύ δραστήριο και η σχέση μας γενικά είναι άριστη. Γι' αυτό υπάρχουν περισσότερες υποθέσεις. Σε μερικού τομεί βέβαια υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά εμένα με ανησυχούν περισσότερο οι χώρες μέλη όπου δεν υπάρχει τέτοιο τόσο λεπτομερές σύστημα παρακολούθησης. Και όπου άρα δεν υπάρχει και τέτοια συνεργασία και τέτοιες ανταλλαγές δεδομένων και άρα και τόσο πολλές υποθέσεις. Για τα Βαλκάνια και ιδιαίτερα τα δυτικά τι αυτά τώρα. Έχουμε κάνει ορισμένες έρευνες στα πλαίσια της προένταξης. Το σημαντικότερο όμως είναι η εκπαίδευση που κάνουμε στην Κροατία, ιδιαίτερα αλλά και σε άλλες χώρες των δυτικών λεγόμενων Βαλκανίων αφιερώνουμε πολύ χρόνο εργασίας του προσωπικού στην επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων από τις χώρες εκείνες για να είμαστε βέβαιοι ότι η επιτήρηση θα γίνει σωστά. Και αυτό θα το συνεχίσουμε και θα το βελτιώσουμε. Η διεθνής αντιαπατική αστυνομία θα αρχίσει να λειτουργεί σε λίγο και λυπάμαι ιδιαίτερα μεταξύ άλλων και γιατί χάθηκε άκερα ο φίλος μου ο Φρανς Μπρούνερ. Ήταν δική του ευθύνη όλα αυτά. Έχουμε στείλει ένα μέλος του προσωπικού μας να παρακολουθεί συνεχώς την Ακαδημία αυτή στη Βιέννη. Τώρα επέστρεψε στις Βρυξέλλες αλλά θα συνεχίσει τη συνεργασία με την Ακαδημία και με μεγάλη συγκίνηση έλαβα ένα γράμμα ευχαριστειών από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας σχετικός. Η συνεργασία με την Ευρωπόλη είναι επίσης σημαντική αν και δεν κάνει την ίδια δουλειά. Εκείνοι συλλέγουν περισσότερο πληροφορίες μόνοι τους και η συνεργασία μας συνεχώς βελτιώνεται. Υπάρχει νέο νομικό καθεστώς με την Ευρωπόλ που επιτρέπει καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων η Όλαφ συμμετέσχε ενεργά σε πολλές δραστηριότητες της Ευρωπόλ η οποία βέβαια καλύπτει πολύ ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Εμάς είναι λιγότερο το μεγάλο το φάσμα και πιο συγκεκριμένο λαθρεμπόριο, τσιγάρων ε, άλλων ειδών χρηματοδότηση της τυρομοκρατίας, τέτοια πράγματα είναι αυτά στα οποία ειδικευόμαστε εμείς σε συνεργασία όμως με την Ευρωπόλ. Υποθετικά τα λέω όλα αυτά, ε, δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Πάντως η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει νέες δυνατότητες και υπάρχουν υποθέσεις που όπου μπορέσαμε να συνεργαστούμε και με τους συναδέλφους μας της Eurojust Τώρα, ο αριθμός των ερευνητών ή των επιθεωρητών. Αν θυμάμαι καλά, 130 είναι περίπου. Αλλά σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό. Υπάρχει προσωπικό που ασχολείται με την τεχνολογία συλλογής πληροφοριών, 85% των υποθέσεων που αφορά είναι συγκεκριμένα της Όλαφ. Έχουμε περίπου 12 ανθρώπους στο λεγόμενο Operational Intelligence Unit και μόνο, αυτοί και μόνο έχουν μεγαλύτερες ηλεκτρονικές δυνατότητες από ολόκληρες κρατικές υπηρεσίες. Έχουμε και ένα τμήμα σήμανσης που χρησιμοποιούμε, αλλά ίσως δεν είναι εδώ το καλύτερο βήμα για να σας τα εξηγήσω όλα αυτά. 75 πάντως της 100 των όρων μας υπολογίζουμε ότι αφιερώνονται σε λειτουργικές δραστηριότητες, στην ερευνητική μας δραστηριότητα και στους τομείς όπου έχουμε αποκλειστική δικαιοδοσία. Αυτά νομίζω κύριε Πρόεδρε είναι αυτά που μπορούσα να πω. Σίγουρα δεν θα απάντησα πλήρω σε όλες τις απαντήσεις, αν χρειαστεί να ξαναμιλήσω. Ο κύριος ναι. Σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά αυτά που είχατε να πείτε κύριε Διευθυντά. Και δημιούργησατε, την εντύπωση ότι οι ερωτήσει μα δεν είναι τόσο καλέ. Γιατί όταν σα πενεύουμε, εμεί λέτε ότι αυτό είναι για τα κράτη-μέλη. Και όταν λέω ότι υπάρχει πρόβλημα, λέτε σωστά. Έχετε δίκιο. Ένα ενίο πρόγραμμα όμως δεν θα λύσει τα προβλήματα. Γιατί όταν έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά την έννοια της απάτης, εσείς αναφερόμαστε πάλι στα κράτη-μέλη, τα οποία το καθένα ορίζει διαφορετικά την έννοια της απάτης. Και όταν βλέπω εδώ στην έκθεση ότι το 2008 68 υποθέσεις ολοκληρώθηκαν. Λέτε εσείς ότι αυτός ο αριθμός είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε μια πιο ευανάγνωση έξω στα χέρια μας για να σας παρακολουθούμε καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω το Διευθυντή αν έχει γνώμη σχετικά με την Κροατία. Διότι ο Πρόεδρος θέλησε να στείλουμε μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας ε, στην Κροατία. Θα μπορούσατε να μας πείτε τη γνώμη σας για το τι γίνεται με τις απάτες στην Κροατία. Είδα ότι έχουμε μόνο μία περίπτωση το 2009. Βλέπουμε στο Βέλγιο έχουμε ένα ψηλό ποσοστό απατών. Τώρα ακούσαμε την εξήγησή σας ότι επειδή έχουμε δηλαδή πολλά θεσμικά όργανα εδώ στις ε, Βρυξέλλες έχουμε και πολλές στατιστικές. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε Δεν θα έπρεπε να αποσυνδέσουμε τις, ε, τα θεσμικά όργανα από το κράτος μέλος ούτως ώστε να μην φαίνεται ότι το Βέλγιο έχει τόσα ψηλά ποσοστά απάτης ο κύριος Ντόιτς. Μάλιστα. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, και εγώ σας ευχαριστώ για την έκθεση και εισήγησή σα. Με βάση την ανταλλαγή αυτή απόψεων που κάναμε έχω δύο σχόλια, δύο ερωτήματα μου γεννήθηκαν. Πρώτον, επανειλημμένος κάθε χρόνο στην έκθεσή σας διαβάζουμε παρατηρήσεις για τις νέες χώρες μέλη. Ερωτώ λοιπόν, στις εκθέσεις της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής ακούγονται ορισμένα στοιχεία, αλλά αυτά τα μαθαίνει η Κομισιόν. Διότι η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια γενική διεύθυνση κατά των απατών και κάνει ορισμένα σχόλια για τις υπηρεσίες που έχει η ίδια συστήσει στα κράτη-μέλη και λέει ότι αυξάνονται έτσι οι κίνδυνοι απάτης αλλά δεν παίρνει υπόψη της στην πράξη τα ίδια της τα σχόλια ή τα σχόλια της Όλαφ αυτό είναι περίεργο. Δεύτερον, εάν η Όλαφ, ρωτώ αν η Όλαφ έχει σκεφτεί καθόλου τη δυνατότητα να αρχίσει κάποιες περιορισμένες έρευνες, όχι πολύ ακριβές, για τον ορισμό της απάτης γιατί υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Και πώς καθορίζεται λοιπόν μέσα στην Ένωση ο ακριβής αριθμός των απατών. Ο αριθμός που δίνουν οι αρχές είναι ένα πράγμα, αλλά υπάρχουν και κρυμμένες, κρυμμένες περιπτώσεις. Τι ποσοστό αποκρύψεως υπάρχει λοιπόν. Για να μπορέσουμε έτσι να δούμε και πόσο αποτελεσματικές είναι οι κρατικές υπηρεσίες διότι οι αριθμοί στις εκθέσεις τη δική σας και της Κομισιόν πρέπει να είναι συγκρίσιμα και να δείχνουν πόσες αποκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχουν. Στο μέλλον δε οι έκθεσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρουν συγκεκριμένα ποια συνεργασία υπάρχει μεταξύ Όλαφ και κρατών μελών. Να κάνετε έναν πίνακα των 27 χωρών που και να κατανέμονται εκεί οι συνεργασίες της Όλαφ με κάθε χώρα μέλος. Με τη Ρουμανία, με τη Βέλγια, με, με όλες. Ένας πίναξ λοιπόν. Πίναξ. Γιατί αυτή τη στιγμή η έκθεσή σας δεν έχει πίνακα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να δίνονται βαθμοί στα κράτη-μέλη, αλλά να παρουσιάζει η Όλαφ τι έχει μάθει, από τι έχει διδαχθεί από τα κράτη-μέλη. Και τρίτον, αν μου το επιτρέπετε, αφού μιλάμε για την απάτη, πρέπει να ξέρουμε ότι κανένας Ευρωπαίος πολίτης δεν αγνοεί τι είναι απάτη από την καθημερινή του ζωή. Είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι οργανισμός καταλαβαίνει ο καθένας τι είναι απάτη. Και εδώ μέσα άμα κοιτάξετε στα πρόσωπά μας θα καταλάβετε ότι κανείς από μας παρά το ότι όλοι γνωρίζουν τι είναι απάτη δεν θα μπορούσε να καταλάβει πώς ακριβώς δουλεύει η Όλαφ και άρα μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς τι συμβαίνει ενώ επαναλαμβάνω καταλαβαίνουμε αυθόρμητα από τα μέσα μας τι είναι απάτη από το μέσα μας και άρα πρέπει οι υπηρεσίες αυτές σαν την όλα που ε, ειδικεύονται στην καταπολέμηση της απάτης να γνωρίζουν τι είναι απάτη. Γνωρίζουν. Χρειάζεται λοιπόν κάποια απλοποίηση των κανονισμών γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ο κύριος Σίλετ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω τι θα ήθελα να πω. Θα πρέπει ίσως να συζητήσουμε διμερώς το θέμα αυτό. Γιατί φοβούμαι ότι δεν σας κατάλαβα απόλυτα και έχω την εντύπωση ότι και εσείς δεν καταλάβετε ακριβώ αυτό που είχα πει εγώ. Ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε λοιπόν διμερώς το θέμα. Για να απαντήσω στον κύριο Ντί. Εγώ ε, Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να κάνω σωστά μία αξιολόγηση της απάντησης στην Κροατία. Πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μία περίπτωση που εξετάζουμε. Αλλά όπως σας είπα, συνεργαζόμαστε στενά με τις κροατικές αρχές για να βελτιώσουμε τις ε, διοικητικές τους ικανότητες και τις ερευνικές τους δυνατότητες. Και ένα από τα προβλήματα που είδαμε να υπάρχει είναι ένα πρόβλημα που είδαμε και σε ορισμένα από τα νέα κρατημέλη. Και στη παλιά κράτη-μέλη ότι το θέμα της ε, δικαιοσύνης ε, δεν ε, προωθείται. Δηλαδή γίνεται μια έρευνα, από την άλλη μεριά όμως το δικαστικό σύστημα δεν μπορεί να παρουσιάσει ένα οριστικό αποτέλεσμα είναι να καταδικάσει κάποιον. Το τελευταίο μήνυμα που μεταβίβασα στις, ε, στις κρατικές αρχές ήταν ακριβώς αυτό, ότι θα πρέπει να εργαστούν περισσότερο πάνω στο θέμα της δικαιοσύνη. Του τουλεχθέντος, εάν θέλετε, μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα briefing πριν από την ε, μετάβασή σας στην ε, Κροατία για να σας βοηθήσουμε αν θέλετε κάτι τέτοιο. Επίσης, η παρατήρηση που κάνατε ε, όσον αφορά τα υψηλά ποσοστά για το Βέλγιο, πραγματικά είναι κάτι που και εμένα ενοχλεί αν πρέπει να το εξηγήσω. Και θέλουμε να το τονίσουμε αυτό στην έκθεσή μας και θα εξετάσω μήπως υπάρχει κάποια δυνατότητα να βελτιώσουμε την παρουσίαση για να μην δίνουμε την εντύπωση ότι πραγματικά το Βέλγιο είναι τόσο πρωταθλητής στις απάτες. θα κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ για να μπορέσω να βελτιώσω αυτό το σημείο. Στρεφόμενο τώρα προ τον κύριο Ντόιτ. για τι εξωτερικέ υπηρεσίε. Πράγματι, δίνουμε χρήσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στην Κομισιόν όσον αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών και συμβάλλουμε σε μεγάλο ποσοστό στην επίλυση των προβλημάτων. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν δεν θέλει να δημιουργήσει περισσότερε υπηρεσίε. Γνωρίζει απόλυτα τις δυσκολίες που υπάρχουν με τις υπηρεσίες αυτές. Όταν υπάρχουν δηλαδή δημιουργίες ε, μικρών σωμάτων εμπειρογνωμόνων, πολλές φορές πολύ μακριά από τις έδρες των θεσμικών οργάνων και περιμένουν αυτά τα μικρά σώματα να σέβονται όλους τους κανόνες και τις διατάξεις που εμείς χρειαζόμαστε πολύ μεγάλο αριθμό ε, προσωπικού για να πετύχουμε. Η πολιτική πραγματικότητα είναι ότι Αυξάνεται ο ρυθμός των υπηρεσιών αυτών όμως από την άλλη μεριά. Και εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής. Και κάτι άλλο θα ήθελα να πω για τις υπηρεσίες. Όταν έχουμε ένα πολύ μικρή σημασία θέμα στην Κομισιόν, που δεν αφορά ίσως απάτη, αλλά κακή συμπεριφορά. προσπαθούν μια ασφαλμένη διαδικασία πρόσληψης. Η Κομισιόν μπορεί να επιβάλλει κάποιε κυρώσει. Οι εξωτερικέ υπηρεσίε δεν έχουν όμω κανένα σύστημα κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή θα εξετάσουμε το θέμα στις ε, υπηρεσίες γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί. Δεν θα το κάνουμε για την Κομισιόν. Και πολλές φορές αποστέλουμε εμπειρογνώμονες στις υπηρεσίες αυτές για να τους βοηθήσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να τους βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε και όσον αφορά το λειτουργικό τμήμα και όσον αφορά το θέμα της ε, πολιτικής για να βοηθήσουμε. Όσον αφορά το θέμα διαφορετικών ορισμών της απάτης, υπάρχει ένα κοινό ορισμός απάτης στα μέσα προστασίας των δημοσιονομικών συμφερόντων των ε, ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Έχουμε δηλαδή ένα κοινό ορισμό και θα πρέπει να θυμούμαστε το θέμα της διαφάνειας και του διεθνούς ορισμού της διαφθοράς που σημαίνει κατάχρηση δημοσίων αρμοδιοτήτων για προσωπικό κέρδος. Αυτή νομίζω είναι ένας καλός ορισμός. Ίσως σήμερα το απόγευμα μακρηγόρησα λίγο για τις δυσκολίες καταμέτρησης. το βασικό επίπεδο απάτης αν θέλετε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία όμως και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί αυτό δεν μπορούμε να το καταμετρήσουμε με τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας στο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε με τις πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας. Η πληροφορία μας είναι καλύτερα όταν α, εξετάζουμε το θέμα των αδασταλιών και όχι τόσο των απατών. Στατιστικά λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε τις πληροφορίες για τα ασθενείς και περνώντας από αυτές να περάσουμε στην στατιστική βάση της απάτης. Αυτό νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια της έκθεσης άρθρο 325 και θα ήθελα ίσως πιο ανεπίσημα και με πιο περισσότερο χρόνο να μπορέσουν να σας ε, παρουσιάσουν το θέμα αυτό οι εμπειρογνώμονές μας, σε όσους ενδιαφέρονται δηλαδή. Και θα ήθελα να περάσω στο επόμενο σημείο του κ. Ντόριτς. Θέλουμε να είναι σαφής η έκθεσή μας όσον αφορά το επίπεδο συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Κανένας δεν μας ε, ε, ζήτησε να έχουμε έναν πίνακα καλών κρατών μελών και κακών κρατών μελών, καλών υπηρεσιών και κακών υπηρεσιών. Αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αλλά δεν είναι αυτή η πρόταση από ό,τι κατάλαβα. Η πρόταση είναι να κάνουμε, για να το πω με δικά μου λόγια, ό,τι μπορούμε για να έχουμε λογικές και πιο λεπτομερείς πληροφορίες προς την κατεύθυνση αυτή να πούμε κάτι παραπάνω στον αφορά το επίπεδο συνεργασία μα με τα κράτη-μέλη, με τι συγκεκριμένε υπηρεσίε, ιδίω ε, να δούμε πού υπάρχει πρόοδο και πού υπάρχουν κενά. Είναι μεγάλο το έργο αυτό και δεν ξέρω ε, τα πόσο θα συστήσω στον επόμενο διευθυντή διευθύντρια για την μελλοντική διευθυνσία έκθεση να το λάβει υπόψη, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη λίγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, πάμε στο επόμενο σημείο. Είναι η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αριθμός 1 κάθετος 2010 και που αφορά στις ε, απλουστευμένες τελωνιακές διαδικασίες εισαγωγής και στον έλεγχό τους. Ο κύριος Στάς, ο εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν γνωρίζω πόσοι διαβάσατε την ειδική αυτή έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά μπορούμε να πούμε ότι το συνέδριο με τους συνεργάτες του έκαναν πολύ καλή δουλειά αξιοσημείωτη και που επιτρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ως προς τις διαδικασίες τελωνιακής απλοποίησης. Είναι πολύ σημαντική η σχετική νομοθεσία για την απλοποίηση των πάντων και του εμπορίου ιδιαίτερα έτσι ώστε οι εμπορευόμενοι να μπορούν πιο εύκολα να, να, να έχουν τις άδειες που χρειάζονται από τις τελωνιακές αρχές. 70% των ε, δοσοληψιών με τα τελωνία βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό καλό είναι καθε αυτόν, καθε αυτό να συνάπτονται συμφωνίες επιλόγω τιμής δηλαδή. Αν γενικευόταν θα ήταν όλα καλά, αλλά απ' την άλλη πρέπει να ξέρουμε ότι πράγματι γίνονται και έλεγχοι και ότι οι συμφωνίες μεταξύ δημοσίων αρχών και των ελεγχομένων ή των ελεγκτικών αρχών ε, είναι σταθερές ώστε το σύστημα να παραμείνει λειτουργικό. Αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν θύλακες απατών, παρακάμψεων, παραβιάσεων της νομοθεσίας και μπορεί ορισμένα ποσά να μην φτάνουν μέχρι τα ταμεία της Ένωσης. Είχα μακρές συνεννοήσεις με μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου στο Στρασβούργο όταν ήμασταν και μετά από αυτές συνέταξα 12 κανόνες, 12 συστάσεις που τη συζήτησα μαζί τους και, και, και, και στην αρχή της ομιλίας του κυρίου Άιλετ συνομίλησα και με άλλα μέλη της Κομισιόν. Έκανα λοιπόν αυτές τις 12 συστάσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη δημοσίευση αυτής της έκθεσης του ηλεκτρικού συνεδρίου γιατί αναγνωρίζω το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι απλοποιημένες αυτές τελωνιακές διαδικασίες αλλά λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί αφού διάβασα την έκθεση διαπιστώνω ότι σημειώθηκαν σημαντικές απώλειες ή θα σημειωθούν για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, για τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Από τις επαφές μου λοιπόν με τους εκπροσώπους της Κομισιόν, που σίγουρα θα ζητήσουν να μιλήσουν σε λίγο, έμαθα ότι και για αυτούς θεωρείται πολύ δύσκολο να κάνουν μια ακριβή αξιολόγηση της σημασίας που έχουν οι απώλειες, αυτές οι ζημίες στον κοινοτικό προϋπολογισμό μετά από, ε, ως αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας ή εφαρμογής των ισχυών των κανονισμών. Έπειτα. Θα ήθελα η Κομισιόν μέχρι τον Μάρτιο του 11, δηλαδή, δηλαδή λέγω τη στιγμή της απαλλαγής, να, να υποβάλει μία βελτιωμένη νομοθεσία πλαίσιο, υπάρχει μεν αλλά βελτιωμένη, ώστε η Κομισιόν να καταλήξει πια, να ολοκληρώσει τις κατευθυντήριες γραμμές που είχε αρχίσει να συντάσει μετά τους πρώτους ελέγχους, διότι ένας από, μία από τις κύριες ελλείψεις στην νομοθεσία μας είναι η έλλειψη συνεργασίας από ορισμένα κράτη-μέλη. Αν δεν συνεργαστούν τα κράτη-μέλη και οι αρχές τους, οι τελωνιακές τους αρχές, αν δεν ασκήσουν τα ίδια τα κράτη τον έλεγχο, ε, τότε η ισχύουσα νομοθεσία δεν εφαρμόζεται ούτε οι συμφωνίες και μπορεί έτσι να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Μπορεί ορισμένοι εγκληματίε να υποφεληθούν από το σύστημα. Επίσης ζητώ στις συστάσεις μου από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν επακριβώς την ισχύουσα νομοθεσία και να φροντίσουν να φροντίσουν να υπάρξει πραγματικός έλεγχος. Η Κομισιόν θα το επιβεβαιώσει αυτό. Θα, θα δούμε ποιοι ακριβώς κάνανε έλεγχο, ποιοι δεν τον κάνανε, ποιοι τον κάνανε περίπου, ποιοι καθόλου κτλ. Και ένα άλλο στοιχείο που συστήνω είναι το 5, δηλαδή, δηλαδή οι πρόσθετες έρευνες και έλεγχοι. Μόλις έμαθα ότι η Κομισιόν πρόκειται στους επόμενους μήνες κράτος το κράτος και συστηματικά να επισκεφθεί επιτόπου τα τελωνία για να δει ποιοι ακριβώς έλεγχοι εφαρμόζονται. Νομίζω ότι θα αρχίσει από τη Δυτική Γερμανία, λέει ο μιλητής, και μετά θα συνεχίσει με την Ολλανδία. Όχι τη Δυτική Γερμανία, την Ομοσπονδιακή Γερμανία. Λοιπόν, πριν καν γίνει η ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού είχαν ανακοινωθεί όλα αυτά και η Κομισιόν πρέπει μέχρι τα τέλη του 11 να έχει μια ιδέα. Ξέρω ότι μέχρι τότε δεν θα τα έχει διαπιστώσει όλα επακριβώς, αλλά μπορεί έτσι η Επιτροπή Ελέγχου του αν έχει στοιχεία για 5-6 ελέγχους, να γνωρίζει περίπου τι συμβαίνει, να έχει μια προσωρινή αξιολόγηση δηλαδή, για να δούμε κι εμείς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και αν υπάρχουν λάθη, παραλήψεις, 25% των πόρων που εισπράττουν τα κράτη-μέλη ως πρόστιμα μπορούν να τα κρατήσουν. Άρα είναι σημαντικό κινητρό αυτό για να κάνουν ελέγχους. Τώρα, για το ελεκτικό συνέδριο του ζητώ να μην παραμείνει σε αυτή την ειδική μονοέκθεση αλλά να παρακολουθήσει, να δώσει και συνέχεια στην ειδική αυτή έκθεση, ώστε να δούμε, ώστε να δούμε λέγω, τι μπορεί ακόμη να βελτιωθεί. Στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, και εδώ είναι η 8η σύστασή μου, προβλέπεται ένα σύστημα ολλανδικό δημοσιονομικού ελέγχου πριν δοθεί κάποια άδεια Θεωρητικά υπάρχει μεν το σύστημα αυτό, η Ολλανδία όμως δεν το εφαρμόζει ακόμα πλήρως. Το θετικό όμως είναι ότι υπήρξε τέτοιο σύστημα και το Ελεκτρικό συνέδριο βρίσκει ότι είναι καλό το σύστημα αυτό. Ζητώ λοιπόν να εξεταστεί πώς θα μπορούσε το πρότυπο αυτό να γενικευτεί ένατη σύσταση για την Κομισιόν αυτή τη φορά. Το σύστημα που λέγεται υπεραπλοποίηση. Θα έπρεπε να δούμε μήπως δεν έχει τύχει καταχρήσεως και αν ναι τι μεγέθους, τι τάξεως. Αυτό θέλαμε να το ξέρουμε πριν την απαλλαγή. Αριθμούς, αριθμούς, αριθμούς. Διότι το σύστημα αυτό της υπεραπλοποίησης κατ' εμέ μπορεί να ανοίξει την πόρτα ή να την έχει ήδη ανοίξει για δημιουργία περισσότερων προβλημάτων. Δέκατη σύσταση. Η Γαλλία, η Ολλανδία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία Εκεί το ερευνητικό συνέδριο διαπίστωσε ότι μερικές επιχειρήσεις δεν ήταν σε θέση να μας δώσουν στοιχεία, τα τελωνιακά στοιχεία που υποχρεούντο να δώσουν. Αν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνουν έρευνες και να φροντίσουμε σε όλες αυτές τις χώρες, όλες, δεν προτιμώ καμία, να γίνει αυτό. Ε, άλλες χώρες που ανέφερε ε, το, το Ελληνικό Συνέδριο τις ανέφερε τις χώρες αυτές. Αυτές λοιπόν πρέπει να εξεταστεί πιο προσεκτικά τι ακριβώς συμβαίνει και η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να γνωρίζει τι, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα των ερευνών αυτών για να δούμε μήπως και το Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να πιέσει. Ο ενδεκάτη σύσταση διαπιστώνω με τα λύπης μου ότι δεν υπάρχει συνεπής πολιτική κυρώσεων. Δεν υπάρχει. Κάθε συμφωνία που παραβιάζεται ή δεν εφαρμόζεται πρέπει να ακολουθείται από κυρώσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε οι κυρώσεις να είναι σοβαρές ώστε τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν τι κίνδυνο διατρέχουν. Και κάτι άλλο που δεν το αναφέραμε, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, διότι εδώ υπάρχει χώρος βελτίωσης. Κάποια επιμόρφωση δηλαδή, να γνωρίζουν και αυτές ποιες είναι οι ευθύνε τους σε περίπτωση μη σεβασμού των διαδικασιών, γιατί άμα το γνωρίζουν αυτό οι επιχειρήσεις, και ε, γίνει επομένως σωστά η εφαρμογή των υπαρχουσών συμφωνιών θα αλλάξουν τα πράγματα. Αν όμως δεν γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους θα καταστραφεί ολόκληρο το σύστημα συμφωνιών συμφωνιών και εμπιστοσύνης και άρα το εμπόριο θα ζημιωθεί. Αυτές είναι οι 12 συστάσεις μου στις οποίες κατέληξα από την εξαιρετική αυτή ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και που ελπίζω να υποστηρίξετε κι εσείς. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Μεσενέ από το ελεγκτικό συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συγγητά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαρστάς για τα σχόλια και τις συστάσεις που διατυπώνει στο έγγραφο εργασίας για την ειδική έκθεση 1-2010 σχετικά με τις απλουστευμένες τελωνιακές διαδικασίες για τις αγωγές. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλο το ιδιαίτερό μου γραφείο και τους συνεργάτες μου στο ελεγκτικό συνέδριο που ε, με βοήθησαν ε, στην έκθεση αυτή. Εγώ διαπιστώνω αυτό το ενδιαφέρον ε, του, της Επιτροπής σας για τη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου για το θέμα αυτό, όπως επίσης και για τα ελλείμματα, τα προβλήματα που διαπίστωσε ο δημοσιονομικός έλεγχος. Λυπούμε όμως που η Κοκομπού τα τελευταία χρόνια δεν εξέφρασε το αντίστοιχο ενδιαφέρον και για τα προβλήματα που διαπίστωσε το ελεγκτικό συνέδριο στον έλεγχο ΝΤΑΣ σχετικά με τα έσοδα του και τα κονδύλια του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν προχώρησε σε ε, ε, ε ή ε, ή τρίλογο μεταξύ της Κοκομπού, της Κομισιόν και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα έλεγα λοιπόν ότι τώρα θα έπρεπε να αναθεωρήσει αυτή τη θέση και να βοηθήσει να έχουμε τέτοιου είδους συνεδριάσεις. Η έκθεση για τις απλουστευμένες τελωνιακές διαδικασίες είναι και η τελευταία έκθεση από πολλές που έχουν ήδη γίνει για το θέμα. Στο παρελθόν το ελεγκτικό συνέδριο εξέτασε το, καθε, το καθεστώς τελωνιακής ε, αποθήκευσης, ε, ε, το θέμα των δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών και το διαμετακομιστικό καθεστώς το 70% των ε, ε, εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008 έγιναν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Επίσης, σε ορισμένα από τα ελεγμένα κράτη-μέλη, οι εισαγωγές με αυτές τις απλουστευμένες διαδικασίες έφτανε στο 93% του συνόλου των εισαγωγών. Χωρίς να είμαι επαναληπτικός, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα θέματα που κατά τη γνώμη του ελεκτικού συνεδρίου αποτελούν κλειδί για τη βελτίωση της ε, τωρινής λειτουργίας των απλουστευμένων τελωνιακών διαδικασιών και που θα εγγυώνται τη σωστή αντίληψη των παραδοσιακών ιδίων πόρων και τον σεβασμό των παραγόγων υποχρεώσεων ε, της εμπορικής ε, πολιτικής της Ένωσης. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι απλουστευμένες διαδικασίες ε, ε, στα τελωνία σημαίνουν ε, γρήγορο, διαδικασίες γρήγορου εκτελωνισμού που σημαίνει δηλαδή ότι ο έμπορος έχει στη διάθεσή του τα εμπορεύματα πολύ πιο γρήγορα σε μικρότερο χρόνο δηλαδή από μια τακτική διαδικασία μειώνονται οι γραφειοκρατίες και οι τελωνιακοί έλεγχοι πριν από την απολευθέρωση δηλαδή των εμπορευμάτων και διευκολύνεται η δραστηριότητα των εμπόρων. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι διαδικασίες αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Το ελεγκτικό συνέδριο ανέλησε τις δύο απλουστευμένες διαδικασίες, τις δύο πιο σημαντικές απλουστευμένες διαδικασίες, είναι η διαδικασία απλουστευμένης δήλωσης και η διαδικασία διαδικασία PDS. Επιτρέπει λοιπόν έτσι να έχουμε σαφείς εγγυήσεις για το πώς γίνονται αντιληπτοί οι παραδοσιακοί ήδη πόροι και ταυτόχρονα σεβόμαστε και τους ε, εμπόρους ε, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έτσι όπως προκύπτουν από τους ε, ευρωπαϊκούς κανόνες. Ανέλησε λοιπόν η το ελεκτικό συνέδριο πώς εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα από τα κράτη-μέλη και από την Κομισιόν. Και θέλησε να διαπιστώσει αν η Κομισιόν εξέτασε σωστά το θέμα του ελέγχου των απλουστευμένων διαδικασμένων, ε, τελωνιακών διαδικασιών και αν επίσης έλαβε υπόψη τις διεθνείς ε, συμφωνίες και την εφαρμογή αυτών των απλουστευμένων διαδικασιών από τα κράτη-μέλη. Επίσης, θέλησαμε να διαπιστώσουμε αν τα εννέα κράτη-μέλη που ελέγξαμε και που αυτά τα εννέα κράτη-μέλη εκπροσωπούν το 60% το 2008 για τους ίδιους πόρους είναι το σωστό παράδειγμα χρήσης των απλουστευμένων διαδικασιών. Και αν ναι, η χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών είναι αποτελεσματική για τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν ε, στην αργοπορημένη της αποτίμηση για την εφαρμογή των μέτρων συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό στα συμπεράσματά της με αυτά του ελεγκτικού συνεδρίου. Βέβαια, ορισμένα, ορισμένες από αυτές τις αποτιμήσεις πρέπει να βελτιωθούν. Πρέπει να εγγυάται η Κομισιόν ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο του 2008 λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ελεγκτικό συνέδριο σύστησε στην Κομισιόν να δημιουργήσει προφίλ, ε, σχήματα ε, στερεότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις, σχετικά με, τις πιο, με τους πιο τρέχοντες κινδύνους και απάτες. Για τα κράτη-μέλη που ελέγξαμε, τα συμπεράσματα του δικαστηρίου λένε ότι δεν γίνονται επαρκείς έλεγχοι διότι δεν υπάρχουν ε, λογικές εγγύησεις για το πώς χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακοί διπόροι. Ούτε κατά πόσο οι χρήστες εφαρμόζουν ε, τις ε, παράγωγες υποχρεώσεις της κοινή εμπορικής πολιτικής. Ο έλεγχος κατέδειξε ότι τα κράτη που ελέγξαμε δεν εφαρμόζουν την ίδια εστίαση του ελέγχου και ότι οι μέθοδοι ελέγχου δεν είναι ε, πάντοτε σωστοί και η έλεγχοι είναι αναποτελεσματική. Διαπίστωσε το δικαστήριο ότι οι εκ των προτέρων ε, έλεγχοι και οι χορηγήσει αδειών ε, για τη χρήση αυτών των διαδικασιών ήταν ανεπαρκής. Ή μετρια, Ήτανε μέτριες. Λοιπόν, ζητήσαμε εμείς ε, να γίνεται έλεγχος αυτών των απλουστεύσεων που διευκολύνουν τους ε, χρήστες και διαπίστωσε ότι υπάρχουν αδικαιολόγητες υπεραπλουστεύσεις. Και επίσης διαπίστωσε ότι δεν γίνονται επαρκείς έλεγχοι εκ ε, των υστέρων. Θέλουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να μηχανογραφήσουν όλες τις απλουστευμένες διαδικασίες. Μαζί με αυτά τα στερεότυπα ε, ρίσκου, τα, προφίλ απάτης, ε, τα οποία επίσης πρέπει να μηχανογραφηθούν. Ολοκληρώνοντας θέλω να ευχαριστήσω και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη δουλειά του κυρίου Μπαρτ και για την, και για την Κομισιόν και να σας πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα προχωρήσει σε ένα follow-up αυτής της ειδική έκθεσης και θα μπορέσει και η Κομισιόν, να, η Επιτροπή σας συγγνώμη, να δει τη συνέχεια των εργασιών της. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τα κράτη-μέλη που θεώρησαν χρήσιμη τη δουλειά μας και πιο συγκεκριμένα τις παρατηρήσεις της Σλοβακίας. Τελειώνω ευχαριστώντας την Επιτροπή σας ε, για, να... για την προσπάθειά της ε, για την πρόθεση της σωστής εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών. Σας ευχαριστώ. Δίνουμε το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς αποτελωνιακής απόψεως να ευχαριστήσω το συνέδριο για την ενδιαφέρουσότατη έκθεσή του. Δεν θα επισέλθω βέβαια σε τόσες λεπτομέρειες γιατί τις κάλυψαν άλλοι. Γενικά νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο και στην εφαρμογή του μπορεί να υπάρξουν ορισμένα στοιχεία που επιδέχονται βελτιώσεως. Γενικά επίσης μπορώ να πω πάλι από τελωνιακής απόψεως ότι δεν έχουμε πολλά προβλήματα και με την έκθεση του κυρίου Στάς του οποίου τις συστάσεις γενικά δεχόμαστε γιατί συμβαδίζουν και με την έκθεσή μας και με τη σφαιρικότερη μας ανάλυση για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα μόνο να τονίσω από δικής μου απόψεως, τελωνιακής δηλαδή, ορισμένα θέματα χρονοδιαγράμματος. Είπε και ο κύριος Στάσης ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε, να επιτηρήσουμε τις χώρες μέλη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είπε ότι θα αρχίσουμε την επίσκεψή μας από τη Γερμανία και μετά την Ολλανδία για να ε, συζητήσουμε εκείνο το την ειδική διαδικασία που εφαρμόζουν οι Ολλανδοί αλλά ίσως χρειαστούν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα γιατί θέλουν, για να έχουμε επισκεφθεί όλες τις χώρες μέλη χρειάζεται πολλή δουλειά και δεν αρκεί μία επίσκεψη γιατί και στο σημείο 3 η έκθεση του κυρίου Στάς μιλάει για κατευθυντήριες γραμμές. Μετά τις επισκέψεις πρέπει να συνταχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές και χρειαζόμαστε κάποιο περιθώριο χρονικό γιατί είναι δύσκολο να γραφτούν οι κατευθυντήριες γραμμές πριν έχουμε επισκεφθεί τουλάχιστον κάποιο σημαντικό αριθμό των χωρών μελών. Αυτό όμως θα το δούμε ίσως διμερώς με το προσωπικό της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τον ίδιο τον κύριο Στάς για να δούμε πώς ακριβώς μπορούν αυτά να διευθετηθούν καλύτερα. Αλλά σαφώς χρειάζεται χρόνος και ο Μάρτιος το 11 είναι πολύ λίγος χρόνος. Ευχαριστώ πολύ. Για το ίδιο θέμα, Πρόεδρε. για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας μας δηλαδή. Και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία του συνεδρίου και την έκθεσή του. Και εμείς παρόμοια προβλήματα έχουμε ταυτίσει κατά τις επισκέψεις μας στις χώρες μέλη. Μάλιστα η Κομισιόν έχει ήδη αναλάβει και δράση και το συνέδριο αναφέρει τους ελέγχους μας που κάναμε το 8 ήδη και χρησιμοποιήσαμε τα συμπεράσματα, τα χρησιμοποίησε και το συνέδριο στην ειδική του έκθεση. Το δε 9 και το 10 η Κομισιόν σε όλα τα κράτη-μέλη διενήργησε τελωνιακούς ελέγχους. Και τώρα συγγράφει μία θεματική έκθεση για τους ελέγχους αυτούς που θα τη συζητήσει προηγουμένως το Δεκέμβριο με εκπροσώπους των χωρών μελών και βέβαια θα το μάθει όλα αυτά και το Κενοβούλιο. Και φέτος θα είναι σημαντικό το θέμα αυτό των ελέγχων και για το αντι-dumping. Για δε το 11 και με βάση τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης θα κάνουμε και άλλους ελέγχους τοπικά για τις τοπικές διαδικασίες συμψήφισης. Και βέβαια πάλι και αυτά θα τα υποβάλουμε στο Κοινοβούλιο. Αλλά έχω και εγώ το ίδιο πρόβλημα με τον προηγούμενο συνάδελφο, το χρονοδιάγραμμα. Δεν προλαβαίνουμε μέχρι το Μάρτιο όλα αυτά προλαβαίνουμε. Ο υπολογισμός τώρα των ζημιών ή απολειών, τι να σας πω, φοβούμαι ότι δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση επ' αυτού ή καμία σίγουρη απάντηση τουλάχιστον διότι η Κομισιόν δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία για να αποφανηθεί Αυτά που μας υποβάλλουν τα κράτη-μέλη είναι πληροφορίες για τα σταλίες και απάτες που έχουν ήδη ταυτίσει. Και οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται στην ετήσια μας έκθεση ή στην έκθεση της Όλαφ που συζητήσαμε στο προηγούμενο σημείο αλλά βέβαια δεν έχουμε πληροφορίες για περιπτώσεις που δεν έχουν ταυτιστεί από τα κράτη-μέλη. Ως Κομισιόν κάνουμε και δικούς μας ελέγχους στα κράτη-μέλη. Αλλά, αλλά το εύρος του δείγματος που μπορούμε να ελέγξουμε είναι πολύ περιορισμένο σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των δοσοληψιών, εκατομμυριών δοσοληψιών. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από όλες. Στους δικούς μας δημοκρατοληπτικούς ελέγχους λοιπόν, οι δοσοληψίες που παληθεύουμε δεν χρησιμεύουν για ποσοτική αξιολόγηση αλλά για ποιοτική για να δούμε αν οι διαδικασίες που ακολουθούν τα κράτη-μέλη και οι αρχές των είναι σωστές. Η Κομισιόν λοιπόν δεν είναι σε θέση να σας κάνει τον υπολογισμό που ζητήσατε. Αλλά να, δεν μπορώ ούτε να σας πω ποιες είναι οι αδυναμίες των διαδικασιών αυτών και που μπορεί να οδηγήσουν ή να οδηγούν σε αδικαιολόγητες απώλειες ή ζημίες γιατί υπάρχουν εκατομμύρια εισαγωγών που δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να τις ελέγξουν όλες. Το σημαντικό είναι το σημαντικό, να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου που να βασίζεται σε σωστή αξιολόγηση ωφέλους κινδύνου για να αποφεύγονται τουλάχιστον οι μεγαλύτερες απώλειες και ζημίες. Πάντως όλα περιορίζονται στις διαπιστώσεις που έχουμε κάνει πράγματι και δεν μπορούμε να ταυτίσουμε παρά επίσημα θα το πω έτσι λάθη όπως λανθασμένα έγγραφα κτλ. Και αυτές όμως οι έρευνες μπορούν να μας δείξουν ότι υπάρχουν μεν αδυναμίες ε, στα συστήματα